Λοιπόν, συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Εξέταση των πράξεων κατεξιοδότηση και των εφαρμοστικών μέτρων. Είναι η 13η φορά που τα εξετάζουμε αυτά. Μια νέα καινοτομία που νομίζω πως είναι σημαντική αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις αρμοδιότητες αυτές του Κοινοβουλίου και οπωσδήποτε η δημόσια συζήτηση είναι βασικό στοιχείο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σήμερα θα ξαναδούμε πάλι την οδηγία για την φερεγγιότητα υπαριθμών 2. Είχαμε τον οργανισμό της 10ης Οκτωβρίου 2014 και την διαδικασία ισοδυναμίας ε, τρίτων χωρών. Και τώρα έχουμε την πράξη κατεξιοδότηση που τροποποιεί τον κανονισμό του 2014 με βασικό στοιχείο η συμπερίληψη μιας ε, κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού υποδομών. Έχουμε τρεις μήνες στη διάθεσή μας να εξετάσουμε αυτά τα πράγματα και μετά τη συζήτηση βλέπετε πως η διαπραγματευτική ομάδα ζήτησε αναβολή και για να εξηγήσει την θέση της διαπραγματευτικής ομάδας θα δώσω λόγο στον κύριο Μπάλτς. και ορίζω και την κυρία Νάταλη Μπερζιέ και τον Τζάστιν Μπρέι στην ΕΙΟΠΑ προϊστάμενο επίσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω σήμερα το πρωί. Να πω κάτι τώρα για τις επενδύσεις υποδομών η Κομισιόν είπαμε δραστηριοποιήθηκε και πρότεινε έτσι μια ειδική κατηγορία στοιχείων ενεργητικού της υποδομές κατά το οποίο οπωσδήποτε υποστηρίζει το ΕΛΚ οπωσδήποτε δεν προλάβαμε να συμπεριληφθεί στο 2015. Βεβαίως η Κομισιόν γνωρίζει τις προθεσμίες Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και μας προξενεί εντύπωση το ότι η Κομισιόν έχει και άλλα σχέδια. Εγώ επιμένω στο ότι η Κομισιόν πρέπει να δημοσιεύσει τα σχέδια αυτά πριν από οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να μας εξηγήσει δηλαδή τι άλλες αλλαγές προβλέπει, τι μορφή θα έχουν αυτές οι αλλαγές πριν περάσουμε το συνολικό πακέτο για την διαδικασία τώρα. Εδώ παρατηρήσαμε ως ΕΛΚ πως ε, η Κομισιόν τα πρότεινε αυτά όλα μαζί ως πακέτο, το λεγόμενο bundling, που είναι προβληματικό, ένα θεσμικό σημείο το οποίο επίσης γνωρίζει η Κομισιόν και είναι σημαντικό για εμάς ως Κοινοβούλιο. Βεβαίω. είναι εξωσημείωτο ότι το νομικό πακέτο πηγαίνει ακόμη ε, παραπέρα καθώς αλλάζουν νομοθετήματα πριν καν εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία. Το ΔΕ Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να εκφραστεί στην κανονική νομοθετική διαδικασία και είναι απλά ε, ένας παρατηρητής. Η ΕΙΟΠΑ Επίσης, μόνο παρατηρητής ήταν και υποθέτω πως η διαδικασία αυτή της διαβούλευσης είναι απλά τυπική και εγώ θα χαιρόμουν ε, αν μπορούσε η Κομισιόν ε, να μας ε, δώσει ακριβώς αυτά τα στοιχεία και κάτι άλλο κάτι το οποίο θα πω ξέροντας πως εγώ είμαι υπέρ της Ένωσης Χρηματαγορών αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να πούμε πως η Κομισιόν έχει μία επιταγή εν λευκό Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το εξής. Όποιος δεν σέβεται την διαδικασία διακινδυνεύει να βρει μπροστά του ένα όχι. Συμπέρασμα. Πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια προγραμματισμού για το μέλλον. Οι ασφαλιστικές ε, εταιρείες ε, στο Solvency 2 σημαίνει πως θα πρέπει να κάνουν ε, τεράστιες αλλαγές και να πάνε από μια ρύθμιση πακέτο σε μια ρύθμιση η οποία θα είναι σταθμισμένη ανάλογα με τον κίνδυνο. Αλλά βεβαίως δεν θα πρέπει να αλλάζουν οι κανόνες κάθε τρεις και λίγο και κυρίως θα μεταλλάζουν τα βασικά τους σημεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να δεχτεί η Κομισιόν να αγνοεί την εντολή των συνομοθετών και να ερμηνεύει την δική της εντολή κατά το δοκούν. Πρόκειται για πράγματα τα οποία έχουν αποφασιστεί εδώ και καιρό και δεν είναι δυνατόν το Κοινοβουλίο να μην ενημερώνεται εγκαίρως για τις προτάσεις αυτές νομοθετικές. Κάτι το οποίο δεν συνέβη αυτή τη φορά, δεν υπήρξε διαβούλευση. Γιατί μόνο αυτό που έγινε δεν μπορούμε να το πούμε διαβούλευση. Δεν είναι δυνατόν το κοινοβούλιο απλά να εγκρίνει ό,τι του σερβίρουν. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω τα εξή ερωτήματα στην Κομισιόν. Πρώτον, πώς θα διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο Δεύτερον, ε, πώς ε, θα μπορέσει να γίνει σε βασούς του Κοινοβουλίου πέρα από τον τριμερή διάλογο. Τρίτον, πώς θα διασφαλίσει η Κομισιόν το ότι δεν θα αλλάζει μια οδηγία πριν καν εφαρμοστεί. Και τελευταία ερώτηση και τέταρτη. Πώς ε, θα ρυθμίσει τις ασφάλειες με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν κάποια στοιχεία να πάνε στον πυλώνα 1 και να μην γίνει καμία σημαντική αλλαγή χωρίς έντολη των συνομοθετών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα νομίζω ότι ναι. η στιγμή να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στη διαπραγματευτική ομάδα. Η Νάταλη Μπερζιέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Γκουαλτιέρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί την απαιτούμενη όθηση για την επίτευξη των στόχων ε, του σχέδιου επενδύσεων για την Ευρώπη και για το σχέδιο περί Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Και οι δύο πρωτοβουλίες έχουν ε, στηριχθεί από το Κοινοβούλιο και ζητήσαμε να κατατεθούν νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να έχουμε μια ε, πλήρως ενοποιημένη Ένωση Αγορών σύντομα για να τονώσουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε τη χρηματοδότηση για να στηριχθούν οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκά έργα. Έχουμε την πράσινη βίβλο για την Ένωση Αγορών από το Φεβρουάριο του 2015. Εκεί προτείνεται, ε, λέγεται μάλλον ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να εντοπιστούν επενδύσεις και ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί και κάποια αναθεώρηση των υποπτικών κανόνων. Ο πρόεδρος Κουαλτιέρη έστειλε και επιστολή το Δεκέμβρη 2014 στον Λόρδο Χίλ μετά την έγκριση ε, του πρώτου κατεξιοδότης κανονισμού Solvency 2 και επίσης υπάρχει ψήφισμα του Ιουλίου 2015 για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών στο οποίο το Κοινοβούλιο τονίζει ότι ε, ένα θετικό περιβάλλον για επιτυχημένη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και για φιλικές οικονομικές, ε, οικονομικούς φιλικούς οικονομικούς όρους. Η ΕΟΠΑ έκτοτε έχει κάνει πολλή δουλειά για τις υποδομές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης ε, για την Ένωση κεφαλαιαγορών καθώς και την παρούσα τροποποίηση κατεξοδότηση πράξης. Σε ό,τι αφορά το γενικό πλαίσιο, οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν ε, ένα περιβάλλον που θα, ε, δεν είναι τόσο ευνοϊκό και γι' αυτό θα πρέπει να διαφοροποιήσουν και να επενδύουν σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που είναι υποφελείς. Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται 10 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία αυτή τη στιγμή. Άρα οποιαδήποτε αλλαγή σε επενδύσεις τους θα μπορούσε να ε, σημάνει σημαντική διαφορά για την οικονομία μας. Ε, η σύγκληση των προτεραιοτήτων δικαιολογεί επιπλέον έργο για το Solvency 2 σε ό,τι αφορά τις κεφαλακές απαιτήσεις με συγκεκριμένε εγγύσει. Το Solvency 2 θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2016. Και δυνάμει Σε ανάληψη αρμοδιοτήτων θα μπορούν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το πλαίσιο πριν το τελικό βήμα. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι να μπορούν να επενδύουν σε project που χρειάζεται η οικονομία μας και ταυτόχρονα να είναι και εποπτικά σωστό το ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε συμβουλή από την ΕΟΠΑ, η οποία ε, μελέτησε τις ε, επενδύσεις σε υποδομές και προέβηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι τροπολογίες εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο και ευθυγραμμίζονται με τις συμβουλές του ΕΙΟΠΑ. Μετά από διαβούλευση της ομάδας εμπειρογνωμόνων ΕΟΠΑ και ΕΚΟΝ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό συμβάλλει τα στο σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιογορών. Αυτή η τροπολογία, η τροποποίηση μάλλον του κανονισμού για την Ένωση Κεφαλαιογορών θεσπίζει μια νέα κατηγορία κινδύνου για τις επενδύσεις σε υποδομές και θεσπίσει συγκεκριμένα κριτήρια που καλύπτουν ε, επιχειρηματικά μοντέλα διακυβέρνηση και εγγυήσει για ένα ευνοϊκό προφίλ ε, κινδύνου. Και δεν περιορίζεται κατηγορία σε οποιονδήποτε τομέα. Απλά επιτρέπει σε καινοτόμα σχέδια τα οποία χρειαζόμαστε να ε, λάβουν τι απαιτούμενε επενδύσει, με λαμβάνοντα υπόψη του στόχου τη στρατηγική του 2020 για μια ανάπτυξη ευφύ για όλους. To non-qualifying investments. Reduce... θα πρέπει να μειωθούν κατά, μειωθεί κατά 40% το τοξικό χρέος και περίπου το, στο 50% ε, το ε, υπόλοιπο χρέο. Αυτή ε, η νέα στάθμιση έχει υπολογιστεί από την ΕΙΟΠΑ ώστε να μετακινηθούν ε, οι επενδύσεις των ασφαλιστών προς επενδύσεις σε υποδομές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται βέβαια υπό τον έλεγχο των ασφαλιστών. Η προληπτική μεταχείριση είναι επιτέλους υγιής και αναλογική εφόσον όλα αυτά λειτουργήσουν ε, ε, σωστά, ε, θα είναι μια πολύ καλή βάση για αυτές τις επενδύσεις. Αυτή η τροπολογία περιλαμβάνει επίσης επιπλέον μέτρα για να υποστηριχθούν οι επενδύσεις στις υποδομές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μία τέτοια ε, προληπτική ε, αντιμετώπιση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα αυτών των ασφαλιστικών εταιριών ε, κατευθύνεται προς τις εταιρείες που χρειάζονται μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Αυτό το μέτρο ακολουθεί τη δημιουργία αυτού του ταμείου μέσω του κανονισμού της 29ης Απριλίου. Αυτό το συγκεκριμένο μέτρο θα ωφεληθεί από τα πιο προσαρμοσμένα ε, ε, ε, τις πιο προσαρμοσμένες κεφαλαιακές χρεώσεις και έτσι αυτή η τελειοποίηση θα επιτρέψει περισσότερο στους ασφαλίστες να επενδύσουν σε προγράμματα υποδομής. Ε, επίσης ε, αυτά όλα διευκολύνονται μέσω των πολυμερών εμπορικών ε, διευκολύνσεων που θα καταγραφούν ως equities γιατί αυτές καλύπτουν από νέους κανόνες μέσω μιας οδηγίας και, ένα κανονισμό, και ενός κανονισμού για τις αγορές και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Επιπλέον η εφαρμογή του μεταβατικού μέτρου που σχετίζεται προς τα equities βελτιώνεται μέσα στο πλαίσιο του, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τους συνομοθέτες, ώστε να αφαιρεθεί οποιοδήποτε κίνητρο για απομάκρυνση των επενδύσεων από τις μικρομεσαίες. Η στάθμιση λαμβάνει υπόψη και τις μη ρευστές equities και θα χαίρει αυτού του πενταετούς προμέτρου του οποίου η εφαρμογή αποσαφηνίζεται για αυτά τα ταμεία. Έχουμε το επίπεδο 1 μεταβατικών μέτρων από το οποίο μετακινηθήκαμε γιατί δεν μπορούσαμε έτσι να καλύψουμε όλο το εύρος του συγκεκριμένου ε, equity. Έτσι λοιπόν είμαστε υπέρ των μικρών και καινοτόμων υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο τόνισε και το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο. Το μέτρο αυτό περιορίζεται στο equity, το οποίο θα αποκτηθεί πριν από την 1η του 16. Ακόμα και αν αυτές οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν ένα περιορισμό, περιορισμένο μερίδιο των 13 του χαρτοφυλακίου μπορούν να σημάνουν τη διαφορά για τις μικρομεσαίες. Τέλος, αυτή η τροποποίηση του εις ε, κατεξιδότηση πράξης Solvency 2 ε, αναμένεται και ε, που δεικνύει πως οι θεσμοί μπορούν έγκαιρα να αντιδράσουν όταν επαρκείς αποδείξεις ε, δείχνουν ότι οι κανόνες μπορούν να βελτιωθούν. Έτσι θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και θα αποφευθεί η απομάκρυση των επενδύσεων από τις μικρομεσαίες, ενώ θα εξασφαλιστεί η προληπτική ε, εξυγίανση ε, όσον αφορά τα επιτόκια. Αυτές οι τροπολογίες ήταν τελευταία ευκαιρία για να ολοκληρωθεί το πλαίσιο του Solvency 2 και η αποτελεσματικότητα των προτάσεων προκύπτει από την έγκαιρη υιοθέτησή του και θα κυρωθεί και θα, από, την, ε, από την έγκαιρη εφαρμογή του. Τώρα βέβαια οι ενδιαφερόμενοι φορείς ε, απαιτούν και αξίζουν ένα προβλέψιμο νομικό περιβάλλον. Η Κομισιόν λοιπόν με, σε βάση αυτές τις προγραμματισμούς και σε, σε ευθυγράμμιση μετά όσα προτείνουν οι συνομοθέτες προ, προτείνουμε την αναθεώρηση στάνταρ που θα ε, διεξαχθεί μέχρι το 2018. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Natalie Berger, now give the floor to Justin Bray. From... Ο Justin Bray από την ΙΟΠΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ΙΟΠΑ καλωσορίζει τις ε, πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε τις κατάλληλες λύσεις για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ταυτόχρονα και όπως τόνισε η Κομισιόν πρέπει το προληπτικό πλαίσιο αυτών των επενδύσεων να αντικατοπτρίζει τους πραγματικούς κινδύνους. Έτσι οι υποδομές ε, μπορούν να εκτιμηθούν καλύτερα από τους ασφαλιστές αλλά ταυτόχρονα πρέπει να τονίσουμε πως τα έργα υποδομών είναι περίπλοκα και απαιτούν μεγάλη εμπειρία. Η Κομισιόν ήδη αναφέρθηκε στις ε, συμβουλές της ε, ΕΙΟΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς ε, της οδηγίας για τη φερικαιότητα Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία είπε η ΕΙΟΠΑ, θα πρέπει να πληρούν κάποιους όρους για την προβλεψιμότητα των ε, χρηματορροών στους επενδυτές, ε, το εύρωστο του πλαισίου και την δυνατότητα να αντέξουν σε κάποια σενάρια κινδύνου. Και βεβαίως ε, ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε το ζήτημα και των αξιογράφων και του χρέους, αλλά προτείνουμε συγκεκριμένα να γίνεται επαρκής δέουσα να ασκείται επαρκής δέουσα επιμέλεια και να γίνονται ναι. σε τακτικά χρονικά διαστήματα stress test όσον αφορά τις ε, χρηματορροές και τη χρηματική αξία των έργων υποδομών. Διαβουλευτήκαμε ευρύτατα, θεωρούμε πως έχουμε αναλύσει το ζήτημα λεπτομερώς και πως αυτά τα οποία λέμε είναι ισορροπημένα και βασίζονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να προσωπήσω εγώ την ομάδα μου, μια που δεν έχει έρθει ο σκιώδης εισηγητής μας. Μετά θα συνεχίσουμε με τις άλλες πολιτικές ομάδες και μετά πάλι ο εισηγητής. Πρέπει να πω πως προσωπικά αλλά και εξ ονόματος των σοσιαλδημοκρατών καλωσορίζουμε αυτή την πράξη κατεξιοδότηση τη ζητήσαμε μάλιστα πρόκειται για μέρος μιας προσπάθειας προσπάθειας να βελτιωθεί ένα μοντέλο που δίνει λανθασμένα κίνητρα και νομίζω πως το να ενθαρρύνουμε τις ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει γιατί ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος γενικά είναι δύο διαφορετικά πράγματα οπότε προσωπικά πρέπει να πω πως εξεπλάγει όταν άκουσα ότι είχε γίνει μια δύσκολη συζήτηση στη διαπραγματευτική ομάδα βεβαίως αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής για το δικαίωμα πληροφόρησης ε, του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό και λυπούμε λίγο για το ότι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, του εισηγητή δεν απαντήθηκαν από την Κομισιόν. Ακούστηκαν κάποια πάρα πολύ καλά επιχειρήματα βεβαίως, όχι ότι δεν απαντήθηκαν αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής. Αλλά το θέμα ήταν το πώς ενημερώθηκε το κοινοβούλιο, κάτι το οποίο για μας είναι σημαντικό, αλλά βεβαίως και η διαβούλευση. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια απογοήτευση για την διαδικασία. Παρόλα αυτά, λόγω της σημασίας της πράξης αυτής εξιοδότηση για την προώθηση των επενδύσεων αυτήν την ΕΛΣΑ και την ΕΛΤΙΦ και τα λοιπά μια προώθηση στην οποία εμείς παίξαμε ένα σημαντικό ρόλο ως κοινοβούλιο νομίζω πως θα πρέπει να σκεφτούμε τα πράγματα προσεκτικά ως κοινοβούλιο για να διακρίνουμε πότε θα πρέπει να ζητήσουμε πλήρη εμπλοκή από τις περιπτώσεις ε, που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν ε, ή να καθυστερήσουν σημαντικά στοιχεία της γενικότερης στρατηγικής μας για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Αυτό ήθελα να πω από πολιτική σκοπιά στην Κομισιόν, την ΙΟΠΑ, αλλά και στην διαπραγματευτική ομάδα. Λοιπόν, ας Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι η δική μου πολιτική ομάδα καλωσορίζει την ευνοϊκή μεταχείριση των, των υποδομών και χαιρόμαστε για την εισαγωγή αυτή ε, αυτών των επενδύσεων στις υποδομές που είναι σημαντικές για την τόνωση της οικονομίας και πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις. Τον προηγούμενο μήνα ζήτησε ε, ε, στοιχεία από την ΕΟΠΑ για τις ε, εταιρείε αυτές. Θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αναλόγως και την κατεξοδότηση πράξη. Θα προχωρήσουμε με προσοχή και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θα πρέπει να αποδεικνύεται, να τεκμηριώνεται. Μας ανησυχεί επίσης ε, η στρεβλωτική συμπεριφορά, αν δοθεί δηλαδή υπερβολική έμφαση σε συγκεκριμένα είδη επενδύσεων, ενώ άλλο όπως για παράδειγμα ε, εταιρικό χρέος ή στέγαση, ε, είναι επίσης οικονομικά βιώσιμε, βιώσιμες κατηγορίες. Θα θέλαμε επίσης ε, η περίοδος κοινοβουλευτικού ελέγχου να παραταθεί για να έχουμε περαιτέρω εξηγήσει από την Κομισιόν για ορισμένα ζητήματα. Θα προτιμούσα να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε την κατεξοδότηση πράξη χωρίς καθυστέρηση. Είναι βέβαια καλό να έχουμε ως σε το δέοντα χρόνο Ελπίζω και να διασκεδαστούν ε, οποιασδήποτε αμφιβολίες και η τροποποιηθήσα πράξη να εκριθεί στο τέλος περίοδου ελέγχου. Ολοκληρώνοντας, έχω ένα ερώτημα προς τους δύο συναδέλφους ΕΟΠΑ και, από την ΕΟΠΑ και από την Κομισιόν. Συγκεκριμένα το ερώτημα είναι, Πέντε χρόνια χρειάστηκε η σχετική νομοθεσία για το Solvency 2 και ταυτόχρονα στο Κοινοβούλιο περάσαμε διάφορες ε, πράξεις για τους οίκους αξιολόγησης ε, και ε, λέγαμε συγκεκριμένα και στο ψήφισμά μας για τα κράτη για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κράτο δεν θα πρέπει να βασίζονται υπερβολικά στις αξιολογήσεις αυτές και νομίζω ότι Υπάρχουν και αναφορές στην νομοθεσία για τις αξιολογήσεις. Οι συνάδελφοι σήμερα το πρωί με πολύ έξυπνο τρόπο απέφυγαν να αναφορούν ε, τις αξιολογήσεις ε, ενώ περίμεναν να αναφέρουν κάτι αλλά κατάφεραν να, μην βάλουν αυτή τη λέξη στις ομιλίες τους. Ε, πώς συμφιλιώνουν όμως ε, την νομοθεσία που έγινε δεκτή για την αξιολόγηση με την ειδική αναφορά στις αξιολογήσεις ε, στη νομοθεσία Solvency 2. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Η Σιλβί Γκουλάρ δεν βλέπω να είναι εδώ. Μαρίζα Ματίας ούτε και αυτή, άρα θα Σβέν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ευπρόσδεκτο το ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε αυτό το θέμα. Και για να βρούμε τα σωστά επιχείρηματα πρέπει να γίνει μια σαφής διάκριση μεταξύ των διατάξεων για τη στήριξη των υποδομών αφενός και αφετέρου της παράτασης about the substance and their arguments about the transitional. Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το equity transition, πρώτα απ' όλα, το δεν το ζητήσαμε, ούτε κανείς άλλος το ζήτησε. Ήταν κάτι λοιπόν που ούτε είχε ε, ζητηθεί από κάποιον. Και τώρα ε, εντάσσονται εδώ και οι μη εγγεγραμμένες, ε, μη συγμένες και από τρίτες χώρες ε, equities ε, μετοχές. Και μιλάμε και για επενδύσεις, όχι για το χρηματιστήριο. Πριν περιοριζόταν εκεί. Εμείς προσπαθήσαμε με να δώσουμε κίνητρα για επενδύσεις που θα γίνονται με αξιόπιστο τρόπο. Και τώρα μιλάμε για μια επέκταση, διεύρυνση επί της ουσίας τώρα. ό,τι αφορά τη διαδικασία και πάλι κάτι για την ουσία όμως. Σε ό,τι αφορά τις κεφαλαϊκέ απαιτήσει, αυτό το λέγουμε calibration, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται ακριβώ. Και η ΕΟΠΑ δεν το έχει απεξεργαστεί νομίζω, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Δηλαδή δεν ήταν ε, στο πλαίσιο της δική σας δουλειά και ούτε, και το αναφέρατε στην παρουσίασή σα Η ΕΟΠΑ λοιπόν έχει εργαστεί πάνω στο calibration, έδωσε σχετικές ε, συμβουλές ό,τι αφορά το equity transitional, διότι εγώ έχω μια διαφορετική εντύπωση για το πώς πήγε η διαδικασία. Υπήρχε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα συζητούσε τις ε, δυνατότητε ε, για τις υποδομές έπειτα. Υπήρχε ένα ευχόλογο από τη Γαλλία που δεν υποστηρίχθηκε από κανένα άλλο κράτο μέλος. Πλήν αγαπητέ μου πρόεδρε της Ιταλίας. Και η Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν υπέρ, κανείς άλλος δεν ήταν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, εν τη σοφία της, το πρόσθεσε το στοιχείο αυτό. συγκεκριμένη κατεξουσιοδότηση πράξη. Και από πλευρά διαδικασία δεν το θέλαμε αυτό. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενεργεί υπέρ θα πρέπει να αφαιρέσει αυτό το, αυτή τη διάταξη. Γιατί διαφοροποιείται από την ε, άποψη της πλειοψηφίας των κρατών μελών, τα είπε Κάσλι Φόξ. Υποδομές. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι από τη δική μας σκοπιά είμαστε υπέρ του να δοθούν κίνητρα στις ασφάλειες για να επενδύουν σε έργα υποδομών. Ευρωπαϊκή Ένωση Αναλογιστών έχει ε, πει ότι αν δούμε από συστημική πλευρά τα πράγματα θεωρούμε ότι πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για την μεγαλύτερη ε, πολυπλοκότητα και, την, λιγό, τα λιγότερα περιθώρια που αφήνουν όλες αυτές, όλες αυτές οι συμβάσεις. Άρα η προσέγγιση της ΕΟΠΑ δεν θα ε, περάσει τα ε, πρότυπα των ε, αναλογιστών, τα αναλογιστικά πρότυπα. Υπάρχουν κίνδυνοι λοιπόν, άρα θα πρέπει τα λάθη βαθμονόμησης, calibration, να σχολιαστούν περισσότερο και οι συστημικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από συστημικού κινδύνου, καταστροφικούς κίνδυνους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι κάτι όμως που δεν το βλέπουμε. Να μελετάτε ε, παρότι έχουμε αυτή τη νέα κατηγορία στον πρότυπο τύπο ή υποδομές έτσι όπως συσχετίζονται. Και τέλο πάντων δεν, τα, δεν θα τα πω όλα, ε, τι λέει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση Αναλογιστών. Μπορείτε να σχολιάσετε την ουσία. Δεν πρόκειται για ε, ε, ριζοσπαστικούς ε, λομπίστες υπέρ των δικαιωμάτων των καταναλωτών πρόκειται για τους που θα πρέπει να τα εφαρμόσουν τα πρότυπα αυτά. Άρα, επί της ουσίας, ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με την κριτική που ασκούν οι αναλογιστέ. Uh, um, I have, uh, now, yes, uh, Danuta Hubner. Ναι, η Danuta Hubner και η Περβάνο Σουμπερές. Μία ερώτηση. Έχω πολίτης δεν έχω εμπλακεί στον κανονισμό αυτόν. Αλλά σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο Σβέν Γκίγκολτ για τη μεταβατική περίοδο. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι με το χικό κεφάλαιο που εκδίδουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνήθως ε, δεν μπαίνει στο χρηματιστήριο και έμαθα από την Κομισιόν πως λέει πως μέσω αυτής της πράξης κατεξιοδότηση αφαιρούν και τα κίνητρα από επένδυσης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς κολλάνε αυτά και γιατί είναι τόσο επικίνδυνο να συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μη εισηγμένες. Μιλάμε μόνο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή γενικά για τις μη εισηγμένες. Το ερώτημα μου είναι προς την Κομισιόν πώς το δικαιολογείτε αυτό. Για να αντιληφθώ θα υποφέρουν, δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τη μεταβατική περίοδο πόσο μεγάλο είναι ο κίνδυνος και πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτά τα κίνητρα από επένδυσης. Ευχαριστώ, Περές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είχαμε μεγάλη ευθύνη καθώς προηγήθηκα ημών στην Προεδρία αυτής της Επιτροπής. Θυμάμαι τις διαπραγματεύσεις για το Solvency 1. Λίγοι είχαν αυτό το προνόμιο εντός της αίθουσας. Ήταν μια μακρά και πολύ ε, βαριά διαδικασία από ένα από τα διακυβεύματα που τονίστηκαν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν ο κίνδυνο να έχουμε ένα επίπεδο 1 το οποίο <coughs> ε, το οποίο εισήγαγε ένα χαρακτηρισμό πολύ βραχυπρόθεσμα και με ένα κατόφλι στις διαπραγματεύσεις σε αντάλλαγμα το άνοιγμα των εσωτερικών αγορών και την επιρροή της σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, και ο ορισμός του κινδύνου α1 ναι. Σύμβουλό σα ήταν η επίση στι διαπραγματεύσει ε, και θα τα θυμάται πολύ καλά και εκείνο. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τη στιγμή όπου ξέσπασε η κρίση στην Ευρώπη, ε, βλέπαμε ποιο κίνδυνο διατρέχαμε μέσα σε αυτό το βραχυπρόθεσμο πλαίσιο. Η εξοδότηση πράξη που προτείνει η Κομισιόν θεωρώ εγώ πως είναι σύμφωνη με τη διόρθωση που αναμένουμε. Με εντυπωσιάζει που ακούω διάφορους συναδέλφους να αναφέρονται σε θέσεις ε, εντός του Συμβουλίου, γιατί είχα την εντύπωση ότι μέσα στην την Επιτροπή είχαμε όλοι υποστηρίξει την ε, το, πόσο, ε, το πόσο λογικό και βάσιμο ήταν το πλάνο Juncker, το σχέδιο Juncker. Δηλαδή, χρειαζόταν να δώσουμε ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις έτσι ώστε τα 315 ε, δις του σχεδίου, εκατομμύρια του σχεδίου Juncker δεν ήταν παρά ένα μήνυμα, ένα σήμα προς την αγορά, προς τις αγορές. Και όταν δούμε ποιοι είναι στην καλύτερη θέση για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη δέσμευση των ιδιωτικών φορέων υπέρ των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, βεβαίω τότε στρεφόμαστε προς τους ασφαλιστέ τι ασφαλιστικέ εταιρείες και έτσι. Η κατεξουσιοδότηση πράξη που προτείνει η Κομισιόν είναι πρόσδεκτη. Αναμένεται δε ως ένα στοιχείο εφαρμογής και συντονισμού των όσων είχε περιγράψει ο Επίτροπος ε, Χίλ ε, στην ε, Ένωση των Κεφαλαγορών και εγώ έχω την εντύπωση πως είναι επίγοντα να στείλουμε στις αγορές αυτό το μήνυμα υπέρ των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και των επενδύσεων στις υποδομές εάν έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή, κάποια τροπολοποίηση ε, ίσως θα έπρεπε να πούμε, να αλλάξουμε μόνο πως αυτός ο ορισμός των υποδομών είναι πολύ περίπλοκος και όχι επαρκώς ε, ευρύς. Αλλά πάντως κάθε μέσο ε, που θα είχε στόχο να καθυστερήσει την εφαρμογή αυτής κατ' εξοδότηση πράξη, θεωρώ πως είναι αντίθετο με αυτό που διαρκώς λέμε σε αυτήν την Επιτροπή. Ξέρω πως έχουμε επιφυλάξει πολλές φορές για τη τάδε ή δίνα πτυχή, ότι δεν μας έχουν διαβουλευτεί αρκετά και ξέρω ποιες είναι οι, και μάλλον λαμβανωμένων υπόψη των θέσεων της Κομισιόν και της ΑΕΟΠΑ δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να είμαστε αντίθετοι. Αντιθέτως θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει όσο γίνεται πιο σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν και η ΕΙΟΠΑ θα μπορούσαν ίσως να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Η Κομισιόν πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Γκουαλτιέρη. Αν μου επιτρέπετε θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, στη σειρά που ετέθησαν. Καταρχήν να απαντήσω στα ερωτήματα του κυρίου Μπάλς. Θα ήθελα να ανανεώσω την δήλωση της Κομισιόν και την προθυμία μας να δηλώσω για την καλύτερη δυνατή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τον εισηγητή. Όσον αφορά και τι μελλοντικέ μας εργασίες, χαρούμε να έχουμε ευκαιρίες για ε, ανταλλαγέ απόψεων. Φυσικά γνωρίζουμε πως αυτή η κατεξουσίδα της είναι ολοκληρωτική στη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αυτό σίγουρα δυστυχώς συνέβαλε σε τμήμα όλης αυτής της βιασύνης και γι' αυτό λυπούμεθα ότι δεν μπορέσαμε δηλαδή να αφιερώσουμε επαρκή χρόνο να κάνουμε αρκετέ επισκέψεις, να το συζητήσουμε διμερώς και να έχουμε και διμερείς διαβουλεύσεις με τον Φυσικά στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι εκτός από την ε, τακτική, την διαβούλευση την οποία κάναμε και όλα στη διάρκεια του καλοκαιριού, εξασφαλίσουμε λοιπόν πως η διαδικασία θα διεξαχθεί όσο γίνεται πιο αμαλά. Για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Φόξ για τη σχέση μεταξύ αυτών, της, της κατεξουσιοδότησης συμπράξης και του κανονισμού για την στάθμιση των οργανισμών. Να τονίσω ότι το Solvency 2 υιοθετήθηκε το 2009, δηλαδή πριν την έγκριση του κανονισμού CRA3 που υιοθετήθηκε στο τέλος του 2012 και βεβαίως ο κανονισμός για τους οργανισμούς πιστοληπτικού πολιτικής ικανότητας ε, ε, συμφωνούσε προς τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν σε επίπεδο G20. Και βεβαίως ε, πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι δεσμεύσεις όπου αυτό γίνεται. Αλλά βεβαίως η παγόρευση έχει στόχο μόνο την αξιοπιστία. Προετοιμάσαμε την κατεξοδότηση πράξη μετά από τις συμβουλές της ΕΙΟΠΑ ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργούσε καμιά μηχανιστική ε, στήριξη για τα οργανισμούς ε, ε, αξιολόγησης. Φυσικά και καταλαβαίνουμε αυτό που εννοείται κύριε Φόξ, αλλά για την ώρα δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το συγκεκριμένο σημείο στο επίπεδο της κατεξοδότησης πράξης. Γιατί εδώ, αν θέλαμε να το κάνουμε αυτό, θα φύγαμε βασικά στοιχεία της νομοθεσίας που έχουν εγκρίνει οι συνομοθέτες. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω μιας πρωτοβουλίας που θα ε, υποβαλόταν σε επίπεδο 1. Και αυτό θα ήταν το τμήμα της γενικής αναθεώρησης που θα γίνει το 2018 Ε, σε σχέση με τον κύριο Γκίγκολτ, κύριο Γκίγκολτ αναφερθήκατε σε κάποιο αίτημα που επέβαλε κάποιο μέλος και που υπευλήθη στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων, όντως ε, είχε υπάρξει ένας κατάλογος μάλιστα αιτημάτων προς τον Λόρδο Χίλ και την Κομισιόν πολύ λεπτομερή αιτήματα, αλλά δεν έχουν ακόμα βρει απάντηση στην κατεξίσου της πράξη και η απάντηση σε αυτά συζητήθηκε στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων και εν γέννη ε, στηρίχθηκε μέσω της ε, στήριξης της πρότασης να γίνει μια αναθεώρηση για να εξεταστούν όλα, αλλά τώρα μέσα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018 πάλι και αυτή η κατεξοδότηση πράξη δεν λαμβάνει υπόψη το αίτημα του κρατών μελών. Αν δει κανεί το μέτρο, και καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε στο συγκεκριμένο μέτρο για το Equity Transitional, θα σας αναφερθώ, θα αναφερθώ σε δύο στοιχεία. Αυτή η πρωτοβουλία παρουσιάζεται σε σχέση με την ε, Ένωση των Κεφαλαγορών και για να αποφύγουμε κινήσεις και απομάκρυνση επενδύσεων που πιστέψαμε ότι μπορεί να συνέβαιναν και γρήγορα, Πρόκειται ένα μέτρο λοιπόν που συνδέεται με αυτό το στόχο και που θέλει να στηρίξει τις επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δεύτερη παρατήρηση επί της οποίας θα ήθελα να επιμείνω είναι ότι πρόκειται μόνο για μεταβατικό μέτρο και ότι είναι μόνο εφαρμοστέο σε ε, equity τα οποία θα έχουν αγοραστεί πριν την 1η 1 του 16. Είναι μεταβατικό μέτρο και ισχύει για maximum 7 χρόνια. Είναι λοιπόν ένα πολύ περιορισμένο μέτρο στην εφαρμογή του και προτείνεται σε σύνδεση με την Ένωση των Κεφαλαίων για να στηριχθούν οι επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, όπως τονίστηκε και από την κυρία Χούμπνερ. Ελπίζω πως αυτή η απάντηση συμβάλλει και στο να απαντήσουμε στο ερώτημα της κυρίας Χούμπνερ, ότι δηλαδή το μέτρο σχεδιάστηκε για να αποφευχθεί ε, το, η απομάκρυνση από τις επενδύσεις και επίσης θεωρήσαμε ότι έπρεπε να, καταγραφ, να ισχύσει για μη ενταγμένες ε, το χρηματιστήριο Equities. Ε, αυτά θέλει να ενθαρρύνει λοιπόν η Ένωση και να τονίσω βέβαια ότι η αλλαγή στο πεδίο εφαρμογή του Transitional ε, θα ωφελήσει όλους τους Ευρωπαίους ασφαλιστές και βασίστηκε σε μια ενίσχυση που δεν περιοριζόταν μόνο στα εγγραμμένα αξιόγραφα. Ευχαριστώ. Η Ιώπα θέλει να προσθέσει κάτι. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω... να σε μια ερώτηση του κυρίου Φόξ και δύο του κυρίου Γκίγκολτ. Ε, την ερώτηση του κυρίου Γκίγκολτ για την αξιολόγηση. Έχει απαντήσει η Κομισιόν, αλλά να απαντήσει και η ΕΙΟΠΑ. Και εμείς βεβαίως γνωρίζουμε την απέτηση που υπάρχει για να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση από τις αξιολογήσεις και γνωρίζουμε πως ειδικά όταν μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα έργα υποδοτών μπορεί να είναι ουσιαστικό το κόστος εξωτερικής αξιολόγησης. Γι' αυτό με έτσι δίνεται η δυνατότητα στα έργα να προχωρήσουν χωρίς αξιολόγηση από οργανισμού αξιολόγησης. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχει η δυνατότητα αυτή και ελπίζω ότι να απάντησα σε ανησυχίες του κυρίου Φόξ. Τώρα, για την ερώτηση του κυρίου Γκίγκολτ για τη μεταβατική περίοδο. Κοιτάξτε, η ΕΟΠΑ απλά παρέχει μια τεχνική προδιαγραφή και άρα να ζητάμε συμβουλές για αυτό το οποίο είπατε για τα αξιόγραφα προ του 2016. Για το τελευταίο σημείο το οποίο αναφέρατε για τις απόψεις των αναλογιστών. Αυτό το οποίο είπατε είναι σωστό. Αν προσθεθεί άλλη μια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού αυξάνεται η πολυπλοκότητα. Αυτό ακριβώς, ε, αυτό είναι το επιχείρημα για το ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειες γιατί αυξάνεται κατά πολύ η πολυπλοκότητα. Μετά όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι Τι σημαίνει αυτό για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού για τις υποδομές. Και νομίζω πως ε, εδώ πέρα τα στοιχεία είναι καλά όσον αφορά το χρέος ε, υποδομών υπάρχει ψηλότερο ποσοστό ανάκτησης ε, αυτού του χρέους σε σχέση γενικά με το εταιρικό χρέος και είναι πιθανότερο να διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του. Και υπάρχουν στοιχεία για το ότι τα αξιόγραφα σε υποδομές ε, αποδίδουν καλύτερα από ότι τα αξιόγραφα γενικώ. Οπότε νομίζω είναι δικαιολογημένο να έχουμε χαμηλές κεφαλιακές απαιτήσεις όταν μιλάμε για έργα υποδομών αρκεί αυτό να συνοδεύεται από στιβαρές απαιτήσει διαχείρισης κινδύνου όπως είπαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως ήταν χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων αυτό το οποίο συζητήσαμε νομίζω δείχνει πως υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω συζητήσεις ε, και διευκρινήσεις μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας και της Κομισιόν. Η πρότασή μου λοιπόν είναι, ενώ λοιπόν α, οπωσδήποτε θα διατηρηθεί αυτό το αίτημα παράτασης ε, να οργανώσουμε αμέσως ε, τις επόμενες ημέρες μία συνάντηση μεταξύ Κομισιόν και Διαπραγματευτικής Ομάδας όπου ελπίζουμε να δοθούν όλες οι διευκρινήσεις όχι μόνο για, το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη πράξη αλλά και για τις ε, επόμενες ε, κινήσεις. Και βεβαίως εάν οι διευκρινήσεις αυτές ε, κρυθούν ικανοποιητικές μπορεί να ξανασκεφτεί το κοινοβούλιο τα διοικητικά του βήματα. Αυτό συμφωνήσαμε με τον Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και αναμένουμε την συνάντηση αυτή το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ τώρα διακόπτουμε για 10 λεπτά μέχρι την ψηφοφορία.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 Dear colleagues, may I ask you to take seat in order to start. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Yes. We start with a test. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Καταρχάς άρχεται η ψηφοφορία. Mm. still a number of colleagues to vote. If you want to test, test. Για να ψηφίσετε όσοι δεν έχετε ψηφίσει ακόμη. Δύο με έχουν, δεν έχουν ακόμη ψηφίσει. Okay. Is, is possible not, not to make the test. It's not mandatory the test. So we close the test. Δεν είναι υποχρεωτικό, λοιπόν. Ξεκινάμε κανονικά να ψηφίζουμε. για την απάντηση εντολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, μυστική ψηφοφορία άρχεται. εγκρίνεται 41 ε, υπέρ 4 κατά 7 αποχές συγχαρητήρι στον κύριο Ενρή. Τώρα παράταση της αιτίας του Προέδρου της ΑΕΟΠ, Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεως Επαγγελματικών Συντάξεων, άρχεται η μυστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται, συγχαίρουμε τον κύριο Μπερναντίνο και τώρα ψηφίζουμε την παράταση της θείας του Προέδρου της ΕΣΜΑ, Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, έρχεται η μυστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Μέιτζορ. Και τώρα περνάμε στην προφορική ερώτηση, σχέδιο προφορικής ερώτησης για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, παράγραφος 1, αρχικό κείμενο, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβιβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, παράγραφος 3, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε τελική ψήφωση. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος για την Ορθίωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Συμβιβαστική B, πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά, άποχες, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία της ομάδας EFTD, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολή 24 έχει αποσυρθεί βαστική C, ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2α, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική D, υπέρ, κατά, ε, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ, κατά, α, έχει αποσυρθεί, συγγνώμη. Όλες δεν το είχα στον κατάλογο. 64 πάμε. Υπέρ, κατά. Και η 43 έχει αποσυρθεί. Εγώ είχα μόνο αυτή ως τις άλλες. Γιατί εξαρτάται από την πολιτική ομάδα που φτιάχνει τον κατά. Τέλος πάντων, η 64 που δεν έχει αποσυρθεί. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε. Ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στην 94. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική λέει ο πρόεδρος 111 Πάμε στα 113. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΆΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το πρόχει 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο στη citation 1, αιτιολογική αναφορά είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε όλες ε, τις, ε, μάλλον μέχρι την 8 όλες ε, τις εντελικές αναφορές υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τώρα από 9 έως και 11, όχι δεν θέλετε, την 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τη 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ετολική αναφορά 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική A, α, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και πηγαίνουμε στα recitals, συντολικές σκέψεις, το α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, α, α μικρό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, το α β μικρό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και σκέψη B τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 έχει αποσυρθεί η 10 δεν έχει αποσυρθεί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο της αιτιολογικής σκέψης B. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Β, α, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο στο C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπω τροποποιήθηκε υπέρ, α, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία.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 εγκρίνεται. 217 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 218 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 219 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο στην πάραφο 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. λεκεί αναφορά citation, α, όλες μαζί, μέχρι τον, ε, την κατηγορία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο recital α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο recital B, Β, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, να ελέγξουμε την τροπολογία 8, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική στο Recital C υπέρ σε δύο τμήματα, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη 17 η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ελέγχουμε τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο recital E κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 και 25 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά. Νομίζω καλύτερα να ελέγξουμε. Θα τα χέρια σας. Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει, δύο. Μάλιστα, πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Συμβαστική Σάιταλ ΕΑ, ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30, υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε άρχεται ψηφοφορία. Την 30. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 32 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική στροσότητα ταλτζή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο Α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 41 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Recital I, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική στο site J, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο site K, K, κατά τμήματα θα ψηφίσουμε. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται M μη σε ένα τμήμα ναι υπέρ να σηκώνω τα χέρια κατά αποχές εγκρίνεται ένα νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Ο όμικρον, όχι. Δύο τμήματα, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της ομικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβεστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρα 22 υπέρ κατά να ελέγξουμε την Ήτρα 22, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Q. Υπέρ. δύο τμήματα μάλλον. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική recital R, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Recital S, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική recital SRA, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο recital T, TAF και εδώ έχουμε ουκολίγα τμήματα. Πρώτον, την προφορική τροπολογία των πρασίνων. Περ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα. Μηματική ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα το έχουν στήσει πράσινη. Πέρα κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε άλλη τμηματική ψηφοφορία. Θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα του αιτήματο των Πρασίνων. Μα ήταν ξεκάθαρο το αποτελέσμα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν δεκτό. Πάμε στο, στην τμηματική ψηφοφορία ECR 8 τμήματα. Υπέρ, το πρώτο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 7. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται το 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 86 υπέρ κατά ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία 86 πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Πάμε στην 100. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 100 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 101. Όχι. Έχουμε πρώτο το αρχικό κείμενο. Το έχουμε, το έχουμε. Υπέρ, κατά, δεν είναι ξεκάθαρο, δεν έχουμε αρχικό κείμενο. Τροπολογία 101, υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται, να το ελέγξουμε όμως. Πέρας. Απορρίπτεται. 122 τροπολογία υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 126. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Τροπολογία 126 με προφορική τροπολογία από τους πρασίνους. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα την τροπολογία χωρίς την προφορική υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την τροπολογία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Ισοψηφία. 27 όλα απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στο U, στη συμβιβαστική για το Essential U,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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 178 με προφορική τροπολογία από την ομάδα Άλντε. Ψηφίζουμε πρώτα την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, άρα το κείμενο της τροπολογίας τώρα ψηφίζουμε υπέρ, κατά, Νομίζω ότι απορρίπτείτε αλλά στο ελέγξουμε, γιατί δεν σηκώσατε τα χέρια αρκετή. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην 200. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το recital W τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική στο X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α1 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 220. Θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, να το ελέγξουμε. Άρχεται ψηφο. Δεν ήσασταν υπέρ. Έτσι νόμιζα. Το δεύτερο της συμβιβαστικής α1. Παράρτημα, άνεξ. Um, Συγγνώμη, δεν υπήρχε δεύτερο τμήμα, γιατί είχε αποσυρθεί η τμηματική ψηφοφορία. Αλλά δεν το είχα εγώ στον καταλογό μου, συγγνώμη, σα ζητώ. Έχει εγκριθεί λοιπόν η συμβιβαστική τελεία. Και πηγαίνουμε στην τροπολογία 220 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ, έχει ψηφοφορία. Vote is Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 224 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται για τη 224. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με την ίδια διαφορά ψήφων. 226 υπέρ, κατά. Ωραία. Πάλι καλό είναι να ελέγξουμε άρχη ψηφοφορία. Μάλλον έχει εγκριθεί βέβαια. Άλλοι δύο να ψηφίσουν. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 232. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη 232 άρχιτη ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Α2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 257 με νέα προφορική τροπολογία από το ΕΛΚ. Η τροπολογία είναι σωμάδα των Δημοκρατών, όμως η προφορική τροπολογία, η καινούργια που λάβουμε είναι από το ΕΛΚ. Λοιπόν, αυτή την τροπολογία την ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρα, περνάμε στη 259 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε τη 259 έρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται συμβιβαστική α4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 282, 282 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 284 υπέρ κατά αποχές νομίζω έχει απορριφθεί να το ελέγξουμε καλύτερα πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται πράγματι 285 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε παρακαλώ έρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική α6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 294. Άρχεται η ψηφοφορία. three colleagues λοιπον περα πέρας. Απορρίπτεται συμβιβαστική α7 σε τέσσερα μέρη. Μέρο πρώτο υπέρ κατά αποχέ δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχέ δεκτό. Τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχέ δεκτό. Τέταρτο μέρο. υπέρ κατά αποχέ δεκτό. 2.98 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 2.98 άρχεται τη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 3.03 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχιε τη ψηφοφορία Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Ε, ήταν ένας παραπάνω, παραπάνω από την άλλη. Δεν πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Όχι, όχι, να ξαναψηφίσουμε, όχι να ψηφίσουμε κατά. Έξι συνάδελφοι ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Άρχισε η ψηφοφορία λοιπόν πέρας και απορρίπτεται με ισοψηφία 312 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 3.13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 418 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τίτλος 1, υπότλος 1 με προφορικές ε, τροπολογίες από τους φάσινους και υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να την επαληθεύσουμε γιατί δεν σηκώνει το χεράκι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β, 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 321 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική β2 α όχι υπάρχει πρώτα η 24 της ήτρα υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία σκεφτεται β Β2 συμβαστική. μέρο πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 351 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Β4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική Β5 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε αλλά ήταν σαφές πέρας αρχικό κείμενο υπέρ κατά Αυτό πρέπει να το επαληθεύσουμε τώρα γιατί κανείς δεν σήκωσε χέρια. Αρχικό κείμενο, τίτλος 2 υπότλο 6, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, τίτλος 2 υπότλο 6, εισαγωγή, υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το επόμενο υπέρ, εδάφιο 1, κατά αποχές δεκτό συμβαστική C1 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική C2 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική C3 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 391 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται απορία Πέρας. Απορρίπτεται. C4. Υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Τροπολογία 401 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 402 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Να το επαληθεύσουμε. 4-0-2 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, είχατε δίκιο, με συγχωρείτε. Λοιπόν, 4-0-3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή συμβιβαστική C7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 412 υπέρ κατά να βαλθεύσουμε την 412 αρχή ψηφοφορία Πέρας. το Αρχικό κείμενο. Unblock. Έχουμε τέσσερα του αρχικού κειμένου. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 4-13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό 4-14 υπέρ μαζί με την 415 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές ε, δεκτό συμβαστική C9 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτό C10 υπέρ κατά αποχές δεκτής D1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 428 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε. Πέραση συμφωρία γκρίνεται 4,29 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την επαληθεύσουμε. ένας παραπάνω από τους πράσινους εξακολουθεί να είναι ένας παραπάνω από τους πράσινους μάλιστα πέρας απορρίπτεται 26 ήτρα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε ή 26, να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Μάλιστα απορρίπτεται. Ή 28, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέτε να το επαληθεύσουμε. Το ίδιο ήταν. Λοιπόν, ψηφίζουμε το κείμενο πώς τροποποιήθηκε. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ναι, άρχεται η ψηφοφορία. και πέρας 45 υπέρ 3 κατά 10 αποχές συγχαρητήρια στους συγητές Now, which one we have to vote now? So, but I need it. Okay. By M.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 Okay, sorry, there was a new problem with. Uh, λοιπόν, συγγνώμη, έχουμε ένα νέο. Νέα ψηφοφορία για την έκθεση BALT. Απολογισμός και προκλήσεις κτλ. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική αλφα. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 30. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΑΒ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 34 ψηφίζουμε Vote is two to vote still. Okay. Vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, όχι 45 γιατί είχε καταπέσει. Α, όχι, 45 υπέρ. Όχι, ναι, μου λένε ότι είναι σωστό. Υπέρ, λοιπόν, ποιοι είναι ότι υπέρ 45 κατά αποχές απορρίπτεται ούτως ή άλλως, αλλά στο ελέγξουμε. Vote is closed. Τέλος της ε, ψηφοφορίας. Απορρίπτεται όντως. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ. Α, σε δύο τμήματα. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική ε, τροπολογία 90, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική μη ε, ε, προφορική από τον εισηγητή μάλιστα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 163 υπέρ κατά αποχές. Ε, α, συγγνώμη, δεν είδα τα χέρια σας. Την νη, την νη ψηφίζουμε. Η μη Μιχάλης συγκρίθηκε. η νη Νίκος ε, την ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά. Ελέγχουμε τώρα την 163. Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 166 υπέρ κατά. όχι, υπέρ, υπέρ, υπέρ, κατά έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον με προφορική των πρασίνων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε τώρα έχουμε το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική π με προφορική του κυρίου Γκίκοντ υπέρ της προφορικής υπέρκατα αποχές ε, απορρίπτεται. Ε, αρχικό κείμενο υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q. Με προφορική ερώτηση των πράσινων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Συμβαστική γιου με χωριστή κατά τμήμα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα Υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Η δεύτερη τμήμα υπέρ αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική χ, x υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική y ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνεται. Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αλφα ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΣ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ΑΔ, AD, με προφορική του κ. Γκίγκολτ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο τη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική ή ε, αε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, τροπολογία 291 υπέρ αποχές ε, απορρίπτεται, η αεφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική ΑΓ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Περκατά κατά αποχές εγκρίνεται, αλφα ε, γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 431 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AJ ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική ΑΚ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική RAL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, συμβιβαστική AM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, AN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σε παράγραφος 33, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 360, 361, 362 είναι ταυτόσιμες. Ε, ποιοι είναι υπέρα ε, κατά έλεγχος ηλεκτρονικός για τις τρεις ίδιες τροπολογίες. Ψηφίζουμε. Νομίζω ότι κρίνονται, αλλά ε, θα το ελέγξουμε τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. δεν ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Περνάμε στο IP ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική αλφακιού. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 377 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, AS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, AT υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΙΟΥ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 490 υπέρ κατά ελέγχουμε την 419 419 Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται ε, αρχικό κείμενο 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ε, αιτιολογική σκέψη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, υπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 2 <coughs> μέχρι 14 έχουμε το αρχικό κείμενο στις αιτιολογικές σκέψεις, έχουμε εγκρίνονται, 3 και 4 είναι ταυτόσημες ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτονται, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνονται, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές ε, ελέγχουμε. Τέλος. W πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική Χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική ΑZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου όπως τοποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. 48 υπέρ, 5 κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ωραία, τώρα ψηφίζουμε... Τίζα, Μόσκα. Οκ. Λοιπόν, σχέδιο γνωμοδότησης για την ΤΙΖΑ. Συμβαστική Α. Χωριστή ψηφοφορία. Μέρος πρώτο. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Να κλείσουμε εδώ αυτή την οθόνη. Ωραία. Μέρος δεύτερο. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μέρος τρίτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική Β. Πρώτα, πρώτα προφορική τροπολογία μάλιστα. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ευσύζουμε το κείμενο ως έχει σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές. Δεκτό, μέρος στο δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την 25 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική A προφορική τροπολογία των πρασίνων υπέρ κατά αποχές απορριπτεται το κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβαστική F υπέρ σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική H υπέρ, μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά Παληθεύσουμε την 65 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε το τελικό κείμενο μοναστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Α, επειδή είναι γνωμοδότηση μάλιστα Πέρας 38 υπέρ 14 κατά 6 αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια τώρα περνάμε στην έκθεση Ρενάτο Σόρου καλά λέω ναι σχέδιο γνωμοδότησης ε, προς μία ενιαία και αγορά συμβαστική α μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές ε, δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε νομίζω ότι απορρίπτεται να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος της συμβαστικής α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική γάμα. Ψήσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά. Να την επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ψηφίζουμε τι συμβαστική έχει υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. τη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές Να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος, άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 44 αρχή τη ψηφοφορία εγκρίνεται συμβαστική ή e, μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος τρίτο υπέρ. Να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος, τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μέρος τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. F. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε η ψηφοφορία. Πέρας. Να απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Να έρχεται η ψηφοφορία. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Α, με συγχωρείτε δεν βλέπω τα χέρια σας πρέπει να την επαληθεύσουμε. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Ποιος εγκρίνεται 91 υπέρ. Κατά να επαληθεύσουμε την 91 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε και αυτήν Πέρας. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά. Α, μα 42 άρχεται η ψηφοφορία, γιατί ζητήθηκε επαλήθευση.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 κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε αρχή ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 121 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 ε, υπέρ. Κατά. Μπορεί να... Δεν ξέρω, μοιάζει διαφορετικά τα πράγματα, να την επαληθεύσουμε. αρχή ψηφοφορία. πέρας δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία του κειμένου όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία πέρας 8 κατά 2 αποχές. Το εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Παπαδημούλη, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Okay, but is I have the, my group, so I prefer yes. to follow this in case you, you, yeah. Okay, we vote the draft opinion. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για την ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το 2014. Εισηγητής ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, συμβιβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γάμα C, η πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής γάμα C. Άρχεται Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται συμβιβαστική δέλτα D με προφορική τροπολογία 2. Δύο προφορικές τροπολογίες. Πρώτη προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, ελέγχουμε, άρχεται ψηφοφορία. Vote is Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 21 προς 27. Δεύτερη προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω καλά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Έρχεται ψηφοφορία. Α, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά τέλος πάντων. Ναι, η ψηφοφορία. Πράγματι απορρίπτεται 21 προς 24. Πάμε στη συμβιβαστική. Συμβαστική D. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. προπολογία 35. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε, ή πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεν βλέπω. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το τμήμα υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε το τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε 45, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πια Τη 47. Να ελέγξουμε τη 47 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 48. Εγκρίνεται. 49. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά δεν ε, βλέπω τους τι κάνουν ελέγχουμε εγκρίνεται φαίνεται μάλιστα τέλος πάντων πέρας ψηφοφορίας ναι εγκρίνεται 52. Συμβιβαστική F, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, άλλο. Να... Μπερδεύκεται, είπα κάτι φώτα. Τέλος πάντων. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Βλέπα κάτι κόκκινα φώτα και είπα ότι απορρίπτεται. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, έτσι ψηφίζαμε. Έληξε ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίφθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική G πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά. Φιλελεύθερη που είναι υπέρ, κατά. Τρίτο τμήμα να ελέγξουμε. Τρίτο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρα ήσασταν κατά εσείς μάλιστα. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πέμπτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε την 65 άρχεται ψηφοφορία Πέρας 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται συμπεριβαστική H, 5 τμήματα, πρώτο, πριν από αυτό, έχω μια προφορική τροπολογία, την οποία θέτω σε ψηφοφόρη από τις Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και τώρα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα, υπέρ,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 απορρίπτεται. Τροπολογία 100 υπέρ, κατά, ελέγχουμε την 100 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε. 107 έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές οι FTD απέχουν απορρίπτεται 111 υπέρ α έχει αποσυρθεί συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική K κατά πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 105 άρχια την ψηφοφορία μάλλον με δύο ψήφους πρέπει να έχει απορριφθεί. απορριφθεί. Τρει συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ναι. Λοιπόν, συμβιβαστική L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική M, μη, πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Η ομάδα SR είναι υπέρ, άρα εγκρίνεται. Εγκρίνεται, ναι. Καλά κάνετε και στη έλεγχο. Πού πάμε τώρα. Τρίτο τμήμα. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική εν, νη. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ο όμικρον, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα 48 υπέρ 5 κατά 4 αποχές συγχαρητήρια στον εισηγητή. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε μια μακρά ώρα ψηφοφοριών. Εγκρίναμε νομίζω σημαντικά κείμενα. Σας ευχαριστώ.